να γίνουν κανονικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δε να προστατευθούν μέχρι την Κυριακή αλλά και μετά την Κυριακή παρατηρητές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα προχωράμε στην έκθεση Μπέλετ, δημόσιες υπηρεσίες ε, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών για το μέλλον, το ψηφιακό μέλλον. Ο εισηγητής έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καλησπέρα σας ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η, Η έκθεση που ελπίζουμε να εγκρίνουμε είναι πολύ σημαντική. Δείχνει μια σοβαρή ε, κατεύθυνση ότι δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει το χαρακτηριστικό ε, μοντέλο μέσων ενημέρωσης που δίνει χώρο και στις ιδιωτικές αλλά και στις κρατικές ε, ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό μοντέλο. Δεν υπάρχει στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία ή βεβαίως στην Κίνα. Το διτό μοντέλο ε, στις περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει δείξει ότι προσφέρει τις καλύτερες εγγυήσεις για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, την ανεξαρτησία των εκδοτών και την ελευθερία του τύπου εν γέννη. Δυστυχώς όμως υφίσταται σοβαρότατες πιέσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης το μοντέλο αυτό, πιέσεις προερχόμενες από διάφορους χώρους. Κράτη-μέλη, όπως επίσης και τις αρμόδιες αρχές, όπως επίσης ε, πίεση από τις ιδιωτικές ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν πίεση στους κρατικούς συναδέλφους. Τους θεωρούν ότι τους ε, υπάρχει αθέμιος ανταγωνισμός μεταξύ τους, κυρίως όσον αφορά τις υπηρεσίες του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσκολεύονται να ορθοποδήσουν. Και αυτό σημαίνει ότι η λεπτή ισορροπία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα διαταράσσεται. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε την επιβίωση αυτού του ε, μοντέλου ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στους δύσκολους καιρούς μας πρέπει να έχει τα μέσα, τα οικονομικά μέσα να επιζήσει στο μέλλον. Ε, αυτό αναφέρει το ψήφισμα. Το πρώτο, και δεν ξέρω αν αυτό είναι πολύ καλά γνωστό, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, δεσμευτεί να προστατεύουν και να εγγυώνται την ελευθερία του τύπου και αναπόσπαστο κομμάτι αυτού είναι το έργο της χρηματοδότησης του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι σαφές και είναι καιρός εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη ότι επιτέλους έχουν ε, αναλάβει τις δεσμεύσεις και πρέπει να τις στηρίσουν. Ένα άλλο θέμα είναι ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης και γενικότερα ελευθερία του τύπου. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας μας. Και γι' αυτό επιθυμούμε ε, να υπάρξει ε, ε, παρατηρητήριο ε, του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης από την Κομισιόν. Είναι πολύ ε, χρήσιμο εργαλείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο προειδοποίησης σε κάποια κρατημέλη ή περιφέρειες όπου η πολυμορφία ε, των μέσων ενημέρωσης και ο πλουραλισμός υφίσταται πιέσεις ή απειλές για πιέσεις. Τέλος δε και πολύ σημαντικό, θεωρώ ότι το σημαντικότερο έργο όλων των μέσων ενημέρωσης στην εποχή μας είναι ε, τα θέματα που έχουν σχέση με το διαδίκτυο. Βλέπουμε όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες στην παρουσία των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στο διαδίκτυο. Κάποιοι συνάδελφοι φαίνεται ότι έχουν ξεχάσει ότι πέρυσι έγιναν σαφείς συμφωνίες και δεσμεύσεις για την δραστηριότητα των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στο διαδίκτυο που πρέπει βέβαια να τηρηθούν. Ως εκ τούτου πρέπει να καθορίσουμε μοντέλα όπου οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών και μηχανών έρευνας πρέπει και αυτοί να παίξουν το ρόλο τους για την ισορροπία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Δεν πρέπει να παραμένουμε αδρανείς γιατί κάποια στιγμή έτσι κι αλλιώς θα ξυπνήσουμε, θα καταλάβουμε το Google, το YouTube και το, Apple έχουν κατακλείσει τον χώρο των μέσων ενημέρωσης, πράγμα που δεν είναι αυτό που επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τρεις συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο με τη διαδικασία διάγει. Ο κ. Μικολάσικ έχει το λόγο πρώτα πρώτα. Πρόεδρε, συνάδελφοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρουμε τη δυνατότητα ισορροπίας παρουσίαση απόψεων, άρα ισορροπίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών αδιοτηλεοπτικών μέσων στην αγορά για να υπάρχει ελευθερία λόγου και να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός. Για την επιτυχία των στόχων αυτών πρέπει να μπορέσουμε να δούμε πώς αντιπροσωπεύονται σε εθνικό επίπεδο και τα δημόσια μέσα. Η ισορροπία μεταξύ εμπορικών και δημόσιων μέσων στα... και στο ίντερνετ πρέπει να είναι βασικός στόχος όλων των πλευρών προς το συμφέρον της αληθούς και σωστής ενημέρωσης. Άλλωστε η ελευθερία των μέσων είναι η βάση της δημοκρατίας. Ο κύριος Χέρενχάουζερ. Ευχαριστώ πολύ. Το, το διτό σύστημα στην Ευρώπη πρέπει να είναι ένα επιτυχημένο σύστημα. Είναι σημαντικό να έχουμε από τη μια μεριά ε, τους δημόσιους και από την άλλη τους ιδιωτικούς ε, ραδιοτηλεπτικούς οργανισμούς, ένα σύστημα ελεύθερης αγοράς. Βέβαια στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι διαφορετικά και βλέπουμε ναι, ότι στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει μια τάση πλήρους ε, μονοπωλίου και αυτή η τάση είναι επικίνδυνη γιατί ε, ε, συμβαίνει σε μια εποχή οικονομικής κρίσης. Από την άλλη πλευρά οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί δεν είναι πάντοτε προσαρμοσμένοι στις ανάγκες και δεν είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς. Και στην Αυστρία ο αντίστοιχος οργανισμός δεν έχει προσαρμοστεί σε αυτά τα οποία θα απαιτούνται σε αυτή την εποχή. Χρειάζεται η πολυφωνία λοιπόν και πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ε, για τη δημιουργία μονοπωλίων είναι κάτι ε, το οποίο εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε φροντίσει πολλές φορές ε, να αναφέρουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροϊτοβά έχει το λόγο. δύο έχουν, θέματα που έχουν σχέση με αυτή τη συζήτηση. Η οδηγία ε, οπτικοακουστικών υπηρεσιών που εγκρίθηκε νωρίτερα βελτιώνει την ε, λειτουργία εποπτείας και επίσης εξασφαλίζει την καλή προστασία των παιδιών από το περιεχόμενο των προγραμμάτων και τη διαφήμιση. Αλλά δεν τηρείται η πειθαρχία αυτή. Δεύτερον, η εναρμόνιση δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να εναρμονίσουμε τον, τον, τρόπο απόκτησης διαμεθοριακών αδειών από όλους τους οργανισμούς. Διαπίστωσα ότι η Κομισιόν πρόκειται του χρόνου να κάνει νέες προτάσεις σε σχέση όμως μόνο με τα έργα μουσικής και όχι με τα οπτικοακουστικά έργα. Θα ήθελα να ρωτήσω πλέον την Κομισιόν να μας πει εάν θα διορθωθεί το θεμελιώδες αυτό λάθος ή Πρέπει εμείς οι Ευρωβουλευτές της Επιτροπές να το κάνουμε. Αυτό ε, μελετά και το άρθρο 33 αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Grazie. La parola all'onorevole Pasca. Ο Πάσκα έχει το λόγο. Πρόεδρε, να υποστηρίξω αυτά που είπε ο εισηγητής, να ανοίξει η συζήτηση για τα μέσα στο Κοινοβούλιο. Το θέμα είναι χρήσιμο, ιδίως τώρα, στην εποχή της ψηφιοποίησης, όταν ε, ο κλάδος αντιμετωπίζει τεράστιες αλλαγές. Ο χώρος των μέσων είναι διαφορετικός. Υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά μέσα. Ε, η σχέση μεταξύ τους ποικίλει από χώρα σε χώρα. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, τα ιδιωτικά μέσα δεν είναι ένα σε άλλες περιπτώσεις είναι και τα μέσα δεν μπορεί να παράσχουν σαφές μήνυμα στους πολίτες. Οι πολιτικές αρχές ωστόσο βλέπουμε ότι συχνά παρεμβαίνουν στην δημόσια τηλεόραση όπου κάνουν οι ιδιώτες για το περιεχόμενο των δικών τους ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης. Πρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία του χρήματος και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης και να απελευθερώσουμε τους ε, δημοσιογράφους για να μην υπόκεινται σε εξωτερικό έλεγχο, αλλά μόνο στον δικό τους αυτοέλεγχο. Διότι αυτοί θα πρέπει να είναι αυτοί που θα αποφασίζουν τι θα παράγουν και αυτή είναι η κύρια αλλαγή που θα πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για την Επιτροπή η κυρία Δαμανάκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, για τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στη ψηφιακή εποχή και το μέλλον του διτού συστήματος. Είναι ένα ισορροπημένο κείμενο το κείμενο της έκθεσης. Υποστηρίζει το διτό σύστημα που βασίζεται στη συνύπαρξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη ραδιοτηλεόραση. Όπως υπενθυμίζει μια αιτιολογική σκέψη η οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα, είναι ένας τομέας που διακρίνει ε, την ευρωπαϊκή ε, αγορά ραδιοτηλεοπτικών μέσων από τις υπόλοιπες αγορές και αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζει η έκθεση το πρωτόκολλο για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη-μέλη αναγνωρίζει την ελευθερία των κρατών μελών ε, να αναθέσουν την εντολή της δημόσιας υπηρεσίας να οργανώσουν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και τη χρηματοδότησή της στο βαθμό που τέτοια χρηματοδότηση δεν επηρεάζει τους εμπορικούς όρους και τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τα κράτη-μέλη καθορίζουν ε, τους όρους χρηματοδότησης ε, των κρατικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων εφόσον τηρούνται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Συμφωνούμε με την ε, βασική γραμμή της έκθεσης ότι τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση και οι νέες πλατφόρμες διανομής σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Αυτό αναγνωρίζεται στην αναθεωρημένη, αναθεωρημένη ανακοίνωση της Επιτροπής του 2009 για την εφαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων ε, στα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Έχουμε ορισμένα σχόλια για δύο σημεία της έκθεσης ε, ιδίως. Καταρχήν όσον αφορά την παρακολούθηση των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, τα, για την ανεξαρτησία των κρατικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων και τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αναθέσουν εντολή στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων χωρίς τη συμφωνία των μελών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, η έκθεση υπονοεί ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν έλαβαν δράσεις για να προωθήσουν ευρωπαϊκά έργα στη ραδιοτηλεόραση. Αυτό δεν υποστηρίζεται από την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής σε σχέση με την οδηγία. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην Ευρώπη πηγαίνουν αρκετά καλά όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα θα πρέπει να βρίσκονται σε ηγετική θέση στην καινοτομία με νέους μορφότυπους και ποιότητα και όσον αφορά το, τα προγράμματά τους και την τεχνολογία για να, να συμβαδίζουν με τις προκλήσεις που τίθενται από παντού. Συμφωνούμε για τα σημεία αυτά και περιμένουμε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά μέσα στο νομικό πλαίσιο που μας παρέχουν οι συνθήκες. Ευχαριστούμε. Περούτε συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη στις 12. Προχωρούμε τώρα στην εξέταση της έκθεσης ΕΛΕΡ πολιτικο-στρατιωτική